Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ καθίστε. Παρακαλώ. Θα αρχίσουμε αμέσως, διότι η σημερινή συνεδρίαση με την παρουσία της Αντιπρόεδρου και της Εκπροσώπου είναι ειδικού χαρακτήρως. Η ημέρη σε διάταξη είναι εξαιρετικά βεβαρημένη. Πρέπει 15 και 45 να κλείσουμε. Παρακαλώ να είστε σύντομοι και ακριβείς. Ο λόγος για τον οποίο συγκεντρωνόμαστε εδώ σήμερα, παρουσία της κυρίας Άστον, αφορά συγκεκριμένα την πολιτική ασφάλειας και άμυνας και δι την ετήσια έκθεση της Υποεπιτροπής, της οποίας έχω την τιμή να προεδρεύω. Σχολιάζουμε λοιπόν την ετήσια έκθεση για την κοινή πολιτική ασφαλείας και άμυνας. Πρόκειται για τις στρατηγικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Πρόκειται για την ε, αναθεώρηση των αμερικανικών προτεραιοτήτων προς τον ειρηνικό, διεθνής ανακρετάξεις και είναι αλήθεια ότι έναντι αυτής της ε, ανακατάταξης η Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές φορές δυσκολεύεται να βρει την θέση της και δει στον τομέα της πολιτικής ασφαλείας και άμυνας. Θα έλεγα λοιπόν ότι η έκθεσή μας είναι μάλλον επικριτική, αλλά απευθυνόμαστε κατά κύριο λόγο στα κράτη-μέλη. Δεν χρειάζεται να παραλάβω, το έχουμε πει τόσες φορές, ότι στον τομέα της άμυνας, στον τομέα των στρατιωτικών, τα κράτη-μέλη έχουν την αρμοδιότητα να λαμβάνουν αποφάσεις. Αυτά λοιπόν πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους ως προς αυτό το οποίο η πλειονότητα των βουλευτών απαιτεί. Σημειώνω επίσης ότι τα θεσμικά όργανα, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, μερικά είναι νεαρά. Χαιρετίζω εδώ τους εκπροσώπους της ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Πολλά λοιπόν από τα θεσμικά μας όργανα δεν είχαν χρόνο να καταφάσκουν στην βούλησή τους ή στην ανάγκη να κάνουμε την παρουσία μας αισθητή Ευρωπαϊκή Ένωση στον κόσμο, στη διεθνή σκηνή. Έχω πολλές ερωτήσεις να θέσω. Θεωρώ όμω ότι όλοι μας θα περιορίσουμε το χρόνο που θα χρειαστούμε. Το ερώτημα που θέτω είναι οι τελευταίες εξελίξεις στο Σαχέλ, διότι εκεί συμβαίνουν οι πιο πρόσφατες εξελίξεις λόγω της επιχείρησης στον Νίγηρα. Έχουμε επίσης την ε, επικείμενη αποστολή στο Μαλί. Είναι θέματα τα οποία έχουμε δείξει λίγο λιγότερο στην εκθεσή μας, διότι πρόκειται για πολύ πρόσφατες εξελίξεις. Αυτά εισαγωγικώς η την πρόσωπος και πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα προτιμήσω να μιλήσω αγγλικά για να είμαι ακριβέστερη. Καταλαβαίνω γαλλικά πολύ καλά, αλλά δυσκολεύομαι πάρα πολύ να μιλήσω γαλλικά όταν ε, μιλώ για θέματα εξωτερικής πολιτικής. Είναι πολύ δύσκολο. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας σας ε, για την ευκαιρία που μου δίνετε να ανταλλάξουμε απόψεις. Είναι πολύ σημαντικό να αφιερώνουμε χρόνο στο να συζητάμε θέματα κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα. Ε, κάναμε τη συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ ε, και ε, το ίδιο επανέλαβα, γιατί αποδίδω μεγάλη σημασία σε αυτά που κάνουμε σε αυτό τον τομέα. Γνωρίζω ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχουν πολλοί υπέρμαχοι του έργου μα και των ευκαιριών των οποίων πρέπει να υποφεληθούμε για να ενισχύσουμε το έργο μα. Την κριτική δεν τη θεωρώ αρνητική. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορείτε ε, να προτείνετε και να επιμένετε σε θέματα όπου θεωρείτε ότι μπορούν να γίνουν περισσότερα πράγματα. Αυτό το οποίο τονίζω είναι ότι όσο περισσότερο συνεργαζόμεθα, τόσο περισσότερο μπορούμε να προωθήσουμε τα σημαντικά θέματα. Οι επιχειρήσεις τις οποίες έχουμε βρίσκονται στο κέντρο της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Και νομίζω ότι μπορούμε να αναφέρουμε συγκεκριμένες δυναμικές εξελίξεις. Έχουμε τις αποστολές στο Σουδάν, στο κέρας της Αφρικής και όπως είπατε εσείς κύριε Πρόεδρε και στο Σαχέλ. Δουλεύουμε ε, για την διαχείριση κρίσεων για δύο δυνητικές νέες αποστολές. Μια στρατιωτική αποστολή στο Μαλί και μια μη στρατιωτική αποστολή στη Λιβύη που θα ασχοληθεί ιδιαίτερα με τη διαχείριση συνόρων, με την ασφάλεια συνόρων. Για να απαντήσω την ερώτησή σας για το Μάλι, ε, στη συνάντηση στις 15 Οκτωβρίου μας ε, ζήτησε το Συμβούλιο να δουλέψουμε πάνω σε μια ε, προοπτική διαχείρισης κρίσεων και αυτό ακριβώς θέλω να παρουσιάσω στους Υπουργού Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνα στο Συμβούλιο της 19 η Νοεμβρίου που θα προεδρεύω. Και μία από τις δυνατότητες τις οποίες ε, εξετάζω είναι να επεκτείνουμε την αποστολή μας EU ε, στα Σαχέλ και Νίγηρα και σε άλλε περιοχέ τη ίδια περιφέρεια. Στου υπουργού εξωτερικών και στου υπουργού άμυνα το έχω αναφέρει πολλέ φορέ και όταν δουλεύω με συναδέλφου που ασχολούνται επιχειρησιακά σε, σε αυτέ τι περιοχέ, το τονίζω πάντοτε ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε το έργο που ξεκινάμε στι αποστολέ μα. Ιδίω ε, έχω κατά νου τη δουλειά που κάνουμε στα Βαλκάνια και όπω γνωρίζετε πολλοί από εσά, πρέπει να το συνδέουμε με τη δουλειά που κάνουμε προσπαθώντα να βρούμε πολιτικέ λύσει. Πιστεύω ότι μπορούμε να υπογραμμίσουμε μερικά πολύ σημαντικά αποτελέσματα που έχουμε επιτύχει και καθοδήγησα την πολιτική μας για την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας ώστε να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Πώς θα γνωρίζουμε ότι επιτύχαμε, τι σημαίνει επιτυχία. Όταν λοιπόν έχω κατά τη δουλειά που κάνουμε στην αποστολή μας στο κέρας της Αφρικής, μπορώ να πω ότι όντως έχουμε σημαντικά αποτελέσματα. Το 2010 ε, ήταν, ε, ε, επλήγησαν από πειρατεία 47 πλοία. Το 2011 μόνο 25 και φέτος το 2012 μόνο 5 πλοία ήταν θύματα πειρατείας. Είναι πάρα πολλά και τα πέντε θα μου πείτε, αλλά η τάση είναι ιδιαίτερα θετική εφόσον μειώνεται. Το 2011 έγιναν 176 επιθέσεις, το 2011 μόνο 35 και μόνο πέντε φέτος το 2012. Και μέχρι τα τέλη του έτους θα έχουμε εκπαιδεύσει 3.000 στρατιώτες, οι οποίοι έχουν συνεισφέρει σημαντικά επιτόπου στη Σομαλία και η κυβέρνηση μπόρεσε να αναλάβει τον έλεγχο μεγάλων τμήματων ε, της επικράτειας της Σομαλίας. Και πήγα μόνη μου στη Σομαλία και είδα τι συμβαίνει επί Συνάντησα τους διοικητές των αποστολών ε, πήγα να συναντήσω τους ε, επικεφαλείς ε, των δυνάμεων εκεί για να συζητήσω μαζί τους πώς βλέπουν εκείνοι την αποστολή και την αποτελεσματικότητα. Υπάρχει λοιπόν όντως επιτυχία. Υπάρχουν βιώσιμα πραγματικά αποτελέσματα. Αυτό όμως που πάντοτε λέω είναι ότι αυτά πρέπει να είναι τμήμα μια ευρύτερη στρατηγική. Και η συνθήκη της Λισαβόνας, ακριβώς αυτή τη δυνατότητα μας έχει δώσει από τη συνθήκη της Λισαβόνας και μετά και χαίρομαι γιατί στην έκθεση επαναλαμβάνεται αυτό το θέμα. Ανέφερε τη Σομαλία και έχουμε επενδύσει πάρα πολλά στο πολιτικό μέτωπο. Και εγώ έχω ασχοληθεί, έχουν ασχοληθεί οι συνάδελφοι επιτόπου, ο ειδικό μα εντεταλμένο Άλεξ Ρόντο. Και όπω σα είπα, επεσκέφθη ε, το Μογκαντήσου τον Αύγουστο και την ε, γύρω περιφέρεια και θεώρησα πολύ σημαντικό να συζητήσω με όλου του διοικητέ των τριών επιχειρήσεών μα ε, για να δω ποια ήταν η γνώμη τους. Και μου μίλησε ο καθένας επαναλαμβάνοντα ότι ήταν, είναι πολύ σημαντικέ αυτέ οι αποστολέ. Είναι ζωτική σημασία στο πλαίσιο μιας γενικότερη προσέγγισης το να σταματήσουμε την πειρατεία στη θάλασσα και παράλληλα να εμποδίσουμε την πειρατεία στην ε, ξηρά. Οι λύσει που θα επιφέρουν ε, το τέλος των συγκρούσεων στη Σομαλία και όταν μιλούσα με τις ε, γυναίκες επιτόπου που ηγούνται των πρωτοβουλειών επιτόπου μου είπαν ότι 30 τόσα χρόνια πραγματικά είναι παραπάνω από αρκετό. Από τότε που ε, υπάρχουν επιτόπου στρατιωτικές δυνάμεις μπόρεσαν να εφαρμόσουν κάποιες ε, ε, αναπτυξιακές ενέργειες που χρειάζεται απαραίτητος η χώρα. Έχουμε συνεργαστεί και με, την, ε, με τους πλειοκτήτες και με τους εταίρους μας όπως το ΝΑΤΟ και την ασπίδα των ωκεανών ε, και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε κατά της πειρατείας και σε συνδυασμό με την αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία. Όταν ε, λέω ότι θα πρέπει να υποφεληθεί ο πληθυσμός της Σομαλίας από όλα αυτά, δεν προσπαθώ να μιλήσω για συμπληρωματικές ενέργειες στην κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, ε, ούτε ε, να μιλήσω μόνο για την ανθρωπιστική βοήθεια. Αντιθέτω, αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να προσδιορίσουμε ένα σωστό μείγμα πολιτικής και τη σωστή διαδοχή των μέτρων και εργαλείων που θα χρησιμοποιήσουμε γιατί έχουμε πάρα πολλά προγράμματα και πρέπει να αντιμετωπίσουμε και την πείνα και την ανάπτυξη ε, και ε, τις βασικές υπηρεσίες ε, εκπαίδευσης και υγείας που πρέπει να παρέχονται. Παράλληλα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν οι εξτρεμιστές και αυτοί που θέλουν να χρησιμοποιήσουν την τρομοκρατία και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όλα αυτά τα οποία πλήττουν αυτές τις περιοχές του κόσμου. Βλέποντας λοιπόν το εύρος ε, των προβλημάτων, καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται μια συνολική προσέγγιση για να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις ανάγκες. Και αυτό που κάνουμε με τις αποστολές της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας είναι ζωτικό ε, τμήμα αυτής της στρατηγικής. Και με αυτό συνδέεται και η πρόληψη και μεσολάβηση των συγκρούσεων. Ε, είμαι ιδιαίτερα ενθουσιώδη για αυτό τον τομέα και ξέρω ότι πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα σε αυτό τον τομέα και αν αποφασίσουμε να έχουμε ένα χωριστό φορέα γι' αυτό θα το υποστηρίξω εφόσον μπορεί να έχει τους κατάλληλους πόρους. Και έχουμε σήμερα την κοινή συνάντηση των Πρωθυπουργών Σερβία και Κωσυφοπεδίου, την οποία θα τους υποδεχτώ ε, και θέλουμε να μπορέσουμε να μεσολαβήσουμε και να μπορέσουμε να παρέχουμε πρόληψη των συγκρούσεων και να βρούμε την υποστήριξη για να μπορούμε να το κάνουμε. Και πάλι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει ένα εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στο να υπάρξει κατανόηση για αυτή την ανάγκη και στο να μας δοθούν οι δυνατότητες να δούμε. Και θέλω να αυξήσουμε τις δυνατότητες μας για να το κάνουμε αυτό και εσωτερικά και εξωτερικά. Αν μου επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να μιλήσω λίγο και για τις δυνατότητε, διότι η κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνας μας δίνει τη δυνατότητα να δράσουμε αλλά πρέπει να έχουμε και τις δυνατότητε για να δράσουμε. Τα κράτη-μέλη δίνουν τις δυνατότητε, και όλοι γνωρίζουμε τις συνέπειες και τι προκλήσεις τη οικονομική κρίση. Γνωρίζουμε τι επιπτώσει στου εθνικού προπολογισμού και στι ε, δυνατότητε Άμυνα και γι' αυτό τονίζω πάρα πολύ ε, την ανάγκη της συνένωσης και κοινή χρήσης. Συνεργαζόμαστε με τους ε, συναδέλφους μας στο ΝΑΤΟ και στα θέματα εφιούς άμυνας και εμείς ακολουθούμε μια διτή προσέγγιση. Καταρχήν έχουμε συγκεκριμένα έργα για τον ανεφοδιασμό εν πτήση. Ένα ε, πολύ σημαντικό θέμα το οποίο ανακαλύψαμε κατά την σύγκρουση στη Λιβύη. Δεύτερον, με την ανάπτυξη της έννοιας της συνένωσης και κοινή χρήσης για να γίνει μια πιο συστηματική προσέγγιση, αυτό θα αποτελέσει ένα τμήμα της εθνικής διαδικασίας προγραμματισμού. Και αυτό θέλουμε να ε, συντεριάζεται αρμονικά με άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές, με την έρευνα και ανάπτυξη, με τη δυτή χρήση, με την αμυντική βιομηχανία με την οποία συνεργαζόμαστε. Όλα αυτά έχουν κέρια σημασία για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά τους πόρους μας. Ε, αυτά και στην έκθεσή σας αναφέρονται κύριε Ντανζόν. Και τα θέματα αυτά είναι στην ημερήσια διάταξη της ε, συνάντησης των Υπουργών Άμυνα στις 19 Νοεμβρίου. Όλα αυτά τα θέματα είναι ζωτικής σημασίας για να είμαστε αποτελεσματικοί. Και ε, θα θέλαμε να είμαστε ακόμη πιο αποτελεσματικοί από ό,τι είμαστε τώρα και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα εξελίσσεται η δουλειά μας μέσα στο παγκόσμιο πλαίσιο Παραδείγματο χάρη, υπάρχει όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον από άλλε χώρε, ιδίω από του εταίρου μα στην Ασία, από την Ινδία, την Ινδονησία, Νότια Κορέα, Βιετνάμ και από την Κίνα, να αρχίσουμε ένα διάλογο για θέματα ασφάλεια και άμυνα. Και όταν πηγαίνω στι χώρε αυτέ, συναντώ του υπουργού άμυνα και εξωτερικών υποθέσεων και προσπαθούμε να εξετάσουμε πώ μπορούμε συγκεκριμένα να συνεργαστούμε. Πρέπει να βασιστούμε σε αυτή την ε, δέσμευση για να είναι τμήμα της στρατηγικής μας να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια σε ολόκληρο τον πλανήτη. Όπως γνωρίζετε, αυτό θέλουμε να συζητηθεί και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και χαίρομαι που ο Πρόεδρος κ. Βαν Ρόμπουι το έχει θέσει στην ημερήσια διάταξη ώστε να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε για τη συζήτηση αυτή στην επόμενη συνάντησή μας τον Νοέμβριο. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να τα εξετάσουμε όλα αυτά μέσα στο σωστό πλαίσιο. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρες οι προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε. Θα πρέπει να είναι σαφές ότι διασφαλίζουμε τους κατάλληλους πόρους για να μπορούμε να δράσουμε και θα πρέπει να είναι σαφές το πλαίσιο μέσα στο οποίο δουλεύουμε. Επίσης, θα πρέπει να είναι σαφές ότι επιτόπου δουλεύουμε ακολουθώντας μία προσέγγιση μακροπρόθεσμη, για να μας φέρει μακροπρόθεσμες και όχι βραχυπρόθεσμες λύσεις. Θέλουμε μια συνολική προσέγγιση. Και θα πρέπει να ε, συγκεντρώσουμε όλα τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, να μπορέσουμε ε, να συγκεντρώσουμε όλους μας τους πόρους και μέσω της Ευρωπαϊκή, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας να αναπτύξουμε ε, νέους τρόπους συνεργασίας, να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία, να υπάρχουν ισχυρές ιδέες για την ανάπτυξη και την καινοτομία, να συνεργαστούμε με ε, τρίτους, με τρίτες χώρες με τις οποίες υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για συγκεκριμένα έργα. Θέλουμε να υπάρχει μια ευρύτερη συνεργασία. Διέτρεξα λοιπόν όλα αυτά τα θέματα για να σας εκθέσω τις απόψεις μου. Θεωρώ ότι πρέπει να προχωρήσουμε και πρέπει να συνεχίσουμε να προωθούμε την έννοια του ότι έχουμε ένα σημαντικό ρόλο να παίξουμε για τη διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας και για τους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για να αντιμετωπίσουμε κάποιες από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ να σας επενθυμίσω ότι είναι πολύ περιορισμένος ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας. Ε, θα σας ζητούσα λοιπόν στις παρεμβάσεις σας να μην ξεπεράσετε το ένα λεπτό. Να επικεντρωθείτε στα θέματα που μας απασχολούν ε, σήμερα. Ξέρω ότι όταν ε, περιβρίσκεται εδώ είπατε εκπρόσωπος θέλετε να αναφέρεστε όχι μόνο σε θέματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική αλλά θα ήθελα να αναφερθείτε στα θέματα που αφορούν την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Σελαφράνκα από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Είπατε πρόσωπα να σας πω ότι από τη δική μας πολιτική ομάδα εκτιμούμε ιδιαίτερα την παρουσία σας εδώ που έχει ως στόχο να βελτιώσει τους μηχανισμούς και της πολιτικής ασφαλείας και άμυνας και αξιολογούμε ότι στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας μας είπατε σήμερα ότι θέλετε και τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εγώ νομίζω ότι εδώ πρέπει να αναζητήσουμε κάποιους τρόπους για να αναπτύξουμε αυτή την καθολική προσέγγιση, την παγκόσμια προσέγγιση προκειμένου να συνδυάσουμε τα διπλωματικά εμπορικά, ανθρωπιστικά και στρατιωτικά μέσα. Και γι' αυτό εγώ νομίζω ότι πρέπει και να επικεντρώσουμε συγκεκριμένε περιορισμένε μέσα και προσπάθειε σε συγκεκριμένε θεματικέ και γεωγραφικέ προτεραιότητε, να έχουμε περιφερειακέ στρατηγικέ μέσα από συγκεκριμένα στρατηγικά έγγραφα. Και πρέπει να ε, όλα, σε τοπικό επίπεδο όλα τα όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση να ασχοληθούν και νομίζω ότι πρέπει να βελτιώσουμε και του μηχανισμού λήψη αποφάσεων και τι εσωτερικέ διαδικασίε για να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα και να δίνουμε γκέρες απαντήσεις. Και κάτι ακόμη Πρόεδρε, συνεργασία με άλλους διεθνούς οργανισμούς, τα Ηνωμένα Έθνη, το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένε Πολιτείε. Στο πλαίσιο αυτό θέλω να ρωτήσω κυρία Άστον, πότε πιστεύετε ότι πέρα από τις συγκεκριμένες δράσεις που μας ανακοινώσετε για το Μάλι, τη Λιβύη, για το κύριο της Αφρικής και τη Σομαλία, πότε πιστεύετε ότι θα κάνετε μια γενική αναθεώρηση σε όλη αυτή τη στρατηγική και ίσως θα ήταν καλό να γίνει το επόμενο έτος ε, όταν θα κάνετε και μια αξιολόγηση της δράσης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας στις εξωτερικές δράσεις. Ευχαριστώ κυρία Γκόμες ε, για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Κυρία Άστον. Ε, είχαμε την τραγωδία του Αμερικανού διπλωμάτη στο Μπεγκάζι. Ε, είναι αλήθεια ότι στη Λιβύη τέτοιες ε, τρομοκρατικές ομάδες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν ε, το κενό που υπάρχει. Όμως μόλις το περασμένο Σαββατό με την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγώ επισκέφθηκα έξω από τον Ζιντάν μια τεράστια αποθήκη πυρομαχικών και ουσιαστικά είναι σαν ένα ανοιχτό σούπερ μάρκετ για τους τρομοκράτες. Εκεί υπάρχουν όλα τα ιδιόπλα από ε, νάρκες κατά προσωπικού ε, μέχρι οποιαδήποτε άλλα όπλα και εκεί ήταν ε, χωρίς να φυλάσσονται, ήταν δεν υπήρχε ασφάλεια. βλέπουμε τι συμβαίνει στο Μαλί και αν ε, τα κράτη-μέλη μας ε, δεν ε, κατανοήσουν ότι πρέπει και η Λιβύη να συμμετέχει στην αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μαλί, τότε ουσιαστικά ε, θα μείνει η κατάσταση ανασφαλής. Ε, δεν μπορούμε να έχουμε ασφάλεια χωρίς τη Λιβύη. Χρειαζόμαστε αυτή τη συνένωση και κοινή χρήση να μεταφραστεί σε δράση. Κατανοείτε ότι τα κράτη-μέλη μας ε, το συνειδητοποιούν αυτό. Σας ευχαριστώ. Κυρία Νέιτς για τους φιλελεύθερους. Καλό σας απόγευμα. Κυρία Στον, αναφέρατε την ε, ανάγκη να αναπτύξουμε στρατηγικό διάλογο με την Κίνα, τη Ρωσία, την Ιαπωνία, την Ινδονησία και να συνεργαστούμε από κοινού για λόγους ασφαλείας. Μία χώρα που δεν αναφέρατε, εκτός αν δεν πρόσεξα εγώ, ήταν η Ρωσία. Και φυσικά η σχέση με τη Ρωσία είναι πάρα πολύ σημαντική και δυσχερής. Υπήρξε πρόσφατη αποπομπή του Υπουργού Άμυνα. Τώρα δεν θα το κρίνουμε εμεί αν αυτό είναι καλό ή κακό. Όμω πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο. Με ρώτησε όμω ένα συνάδελφο που ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το θέμα αυτό και ορθώ. Τι σκοπεύετε να κάνετε για τη σύσταση που ενέκρινε το Νοέμβριο στο Στρασβούργο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με τον επιβάλλη τουλάχιστον περιορισμού στις θεωρήσεις σε όσους είναι υπεύθυνοι για το θάνατο του κ. Μακνίσκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μπράτνερ. Κυρία Άστον, χαίρομαι για την έμφαση στην συνολική προσέγγιση. Και αδελφός μου Συμφώνησε. Χαίρομαι για όλα αυτά. Εντάχει για το Μαλή. Ακούσαμε πολλά. Ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε την Αλκάιντα και άλλε συναφείς οργανώσεις. Όμως υπάρχει και η αντιπολίτευση των Τουαρέγ. Κάποιοι συντάσσονται με την Αλκάιντα, αλλά κάποιοι έχουν αναθεωρήσει. Τι θα κάνουμε αν επέμβουμε στρατιωτικώς, για να μην επιστρέψουν στους συμμάχους στη λάθος πλευρά. Είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε σχέδιο σε αυτή την περίπτωση. Και επίσης για το κοσυφοπαίδιο, το ελεγκτικό συνεδρίο πήγε στην περιοχή και συνιστούν ότι χρειάζεται να ενισχύσουμε τις δυνατότητες μας στην περιοχή. Τι λέτε γι' αυτό. Και για τις δυνατότητες το πολίτε, δημοσιονομικό πλαίσιο μειώθηκε ήδη για εμά τουλάχιστον κατά 10%. Η υψηλότερη μείωση σε σύγκριση με κάθε άλλο τομέα. Πληττόμεθα εμεί, η εξωτερική πολιτική, η ασφάλεια. Τι θα κάνετε γι' αυτό. Και όσον αφορά τι ικανότητε διαμεσολάβηση, είπε όπου δεν μπορούμε να το κάνουμε εσωτερικά, να το κάνουμε σε συνεργασία με εξωτερικού φορεί. Πώ θα γίνει αυτό, κύριε Λόζινγκ. Κύριε Λέζον, ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θα ήθελα να συμφωνήσω και εγώ με αυτά που είπε η συνάδελφος, κυρία Πάρτνερ, ότι χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα για το Μάλι. Από το Μαλί μου λένε ότι Υπάρχουν διάφορε ευκαιρίε διαπραγμάτευση, τις οποίες θα έπρεπε να εκμεταλλευτούμε για διαπραγματεύσεις με τις διάφορες ομάδες των ΑΡΕΓ. Περισσότερο θα ήθελα να αναφερθώ στις στρατιωτικέ πτυχές και να αναφερθώ σε κάτι το ανέφερε ο Χάραλ ε, Κούιεκ, γενικός στρατιωτικό εκθεωρητή. Είχε πει ότι υπάρχει ένα στρατό των 2.000 ατόμων μόνο και θα έπρεπε να εξετάσουμε καλύτερα τις προοπτικές ανάπτυξης επιτόπου θα έπρεπε ενεργά να ασχοληθούμε με την ε, ε, βοήθεια επιτόπου. Θα ήθελα λοιπόν να σας ε, ρωτήσω συγκεκριμένα αν συμφωνείτε με την άποψη του κυρίου Κούγιακ και αν έχετε κάποιο πρόγραμμα, τι πρόγραμμα έχετε για την ανάπτυξη δυνάμεων επιτόπου και τι προοπτικές βλέπετε να δράσετε λίγο πιο αποφασιστικά από αυτό που ήδη μας αναφέρατε. Ευχαριστώ. Ο των έκλεισε. Έχουμε άλλους τέσσερις ομιλητές. Συντομότητα, παρακαλώ. Ο κ. Τζένης, ε, σκιώδηση της για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι παρατηρήσει μου είναι πιο γενικού χαρακτήρα. Γιατί πολύ πρόσφατα συζητήσαμε και την έκθεση Ναντζάν. Σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στα πλαίσια της κοινή πολιτικής ασφαλείας και άμυνας έχουν κάνει μία δήλωση αρχής. Εγώ υποθέτω ότι υπάρχει μία ε, ευρύτερη συμφωνία πέρα από το δικοματισμό, αυτό το κοινοβούλιο είναι υπέρ μία τέτοιας πολιτικής υπάρχουν ε, πάρα πολλοί που αντιτίθεται στο να ε, διαδραματίσει η Ευρώπη, ε, να διαδραματίσει η Ευρώπη ένα πρωταγωνιστικό ρόλο παγκόσμια. Όμως, καθώς βλέπω εδώ τον κύριο Νταντζέν, εγώ θα ήθελα να φτάσω λίγο πιο μακριά στην παρέμβασή μου. Θέλω να ρωτήσω την κυρία Άστον, η διαδικασία που ανακοινώθηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε σχέση με την ε, συγχώνευση ε, της ads ε και της Van System δεν υπήρξε καμία εξήγηση σε σχέση με το θέμα αυτό, αλλά εγώ θα ήθελα να μου πείτε αν εσείς ήσασταν υπέρ μιας τέτοιας συγχώνευσης των μεγάλων ευρωπαϊκών συστημάτων ή όχι. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Κοπά. Ευχαριστώ πολύ. Την περασμένη εβδομάδα επισκεφθήκαμε το Σερβικό Κόσοβο, ταυτόχρονα σχεδόν με την Υπουργό Εξωτερικών Κλίντον, η οποία επισκεφτόταν την περιοχή. Κατά τη διάρκεια της επισκεψεώς μας διασχίσαμε τα βόρεια του Κοσφοπεδίου συναντήθηκα με την Γιούλεξ η οποία μα ενημέρωσε για την κατάσταση επιτόπου. Και παρά την ευγενική διατύπωση αισθανθήκαμε ότι είναι μάλλον ε, απογοητευμένη η αξιωματική τη K4, όχι τόσο λόγω τη έλλειψη συντονισμού επιτόπου όπω λέγεται στην εκθεσή Ντανζό. αλλά για την αδυναμία τη Γιούλεξ να εκτελέσει τα καθηκοντά τη χωρί την υποστήριξη των δυνάμεων του ΝΑΤΟ. Και αυτό επιβεβαιώθηκε από την Ulex. Ως πιθανή λύση θα μπορούσε και η k να συμπληρωθεί με αποστολή ΚΠΑ. Πιστεύετε, είπατε εκπρόσωπο, ότι η ιδέα αυτή μπορεί να υλοποιηθεί. Είναι κάτι που έχει συζητηθεί στο Συμβούλιο, έχει ανταλλάξει υπόψη, ανταπόψη ενδεχομένω από αυτού του θέματο με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Ευχαριστώ, κύριο Σκάτσίν. Πρόεδρε κυρία Θα συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε η κυρία Κοπά και θα πω δύο λόγια για τη σχέση μεταξύ Σερβίας και Κωσοπεδίου. Θέλω να σας συγχαρώ για όλα όσα έχετε πετύχει ως σήμερα. Οι πρόεδροι θα έρθουν στο Μοντενέγκρο, θα συνεχίσετε μαζί τους. Όμως λόγω της ε, απουσίας διαλόγου μεταξύ Βελγραδίου και Πριστίνα επί ο διάλογος ε, γίνεται εσωτερικά μεταξύ Σέρβων του Κοσμοπεδίου. Οι Σέρβοι του ποταμού Ήμπαρ αναγνωρίζονται ως σχεδόν προδότες. Πρέπει όμως αυτό να το καταλάβει το Βελιγράδι. Γι' αυτό ειλικρινώς προτείνω να οργανωθεί συνάντηση μεταξύ του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης του Κοσμοπεδίου και ενός εκ των Αντιπροέδρων στο Βελιγράδι. Αυτό θα είναι πιστεύω πραγματικά μια νέα γέφυρα, ένα νέο βήμα προς τα εμπρός, άμεσος διάλογος δηλαδή μεταξύ των Σέρβων βορείας του Κωσόβου και των Σέρβων που μένουν σε θύλακες και οι οποίοι να συμμετέχουν στην κυβέρνηση. Ευχαριστώ κύριο Στάνοκ. Ευχαριστώ θα μπορούσα να ρωτήσω για τη Συρία, για το Ιράν και για πολλά άλλα θέματα, αλλά θα σας θέσω μία απλή ερώτηση. Ποιος θα αντικαταστήσει ε, την κυρία Κλίντον ως Υπουργός Εξωτερικών. Έχετε κάποια πληροφορία, κυρία Λούνατσεκ. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Βαρονιά Άστον που παρευρίσκεται εδώ και επίσης ε, θα συνεχίσω τα όσα είπαν η κυρία Κοπά και ο κύριος Κατσίνη. Ήμασταν μαζί σε αυτή την επίσκεψη στην Πριστινά και στο Βελιγράδι, το πρώτο κοσυφοπαίδιο, λίγο πριν φτάσατε εσείς με την κυρία Κλίντον ε, και θέλω να σας συγχαρώ. Ε, επειδή καταφέρατε να συναντηθούν οι δύο πρωθυπουργοί και ελπίζω να συνεχιστεί αυτή η επικοινωνία με το απαραίτητο αποτέλεσμα. Η αποστολή Γιούλεξ και η έκθεση του λεκτικού συνεδρίου της περσμένης εβδομάδας, η έκθεση ασκούσε κριτική για την κατάσταση στο Κωσυφοπέδιο, αλλά ασκούσε και κριτική για το πώς διαχειρίζεται την κρίση η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο συντονισμός μεταξύ της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης και των κρατών μελών για τη διασφάλιση λόγου χάρη ότι ε, υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό για τον κατάλληλο χρόνο και έχει τα απαραίτητα προσόντα. Επίσης, ότι οι πέντε κράτη-μέλη δεν έχουν ε, αναγνωρίσει ε, το Αυτό βλάπτει τη δράση της Γιούλεξ. Και επίσης, το γραφείο στην Πριστίνα δεν έχει το απαιτούμενο προσωπικό για να παρουσιάσει τα απαιτούμενα αποτελέσματα. Έτσι, λοιπόν, πώς θα δώσετε συνέχεια σε αυτές τις τάσει του λεκτικού συνεδρίου για να είναι επιτυχές και κάτι να ρωτήσω για τη συμμετοχή των γυναικών εικόνε, στι μη στρατιωτικέ αποστολέ, όχι μόνο στη Γιουλέξ, γενικά τι επιτυχίε είχατε, αλλά και τι πρέπει να γίνει ακόμη και τι δράση να λαμβάνετε. Ευχαριστώ, κυρία Άστον. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλου του ομιλητέ για τι ερωτήσει του και θα προσπαθήσω να απαντήσω στο δυνατόν πληρέστερα. Ο κύριο Σαλαφράγκα Αναφέρθηκε στην συνολική προσέγγιση που θέλουμε να περιλαμβάνει και το διπλωματικό στοιχείο και το εμπορικό και το εκπαιδευτικό στοιχείο. Θέλουμε να είμαστε περισσότερο αποτελεσματικοί στο πώς ε, μπορούμε να προωθήσουμε ε, αυτή την ενιαία δράση και τι ευκαιρίες έχουμε. Πιστεύω ότι είναι πολύ καλή αυτή η ιδέα και για μένα αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι αυτό που κάνουμε μετά τη Λισαβόνα βλέπουμε τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και τι καινούριο μπορούμε να κάνουμε. Βλέπουμε όλους τους διαφορετικούς τρόπους ε, με τους οποίους δράσει ολόκληρο τον κόσμο η Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουμε να έχουμε ένα συνδυασμό στοιχείων που θα μας βοηθήσει μακροπρόθεσμα κάθε στοιχείο είναι ζωτική σημασία από μόνο του. Χρειαζόμαστε ανθρωπιστική βοήθεια για να βοηθήσουμε του ανθρώπου επιτόπου Χρειαζόμαστε αποστολέ τη κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα για να αντιμετωπίσουμε του κινδύνου. Χρειαζόμαστε κατάρτιση και εκπαίδευση προσωπικού. Χρειαζόμαστε ανθρώπου επιτόπου σε πολλέ άλλε περιπτώσει. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Αλλά όχι από μόνο του το καθένα. Δεν θα μπορέσουν από μόνο του το καθένα αυτά τα στοιχεία να εκπληρώσουν αυτά τα οποία θέλουμε. Η συνολική τους ανάπτυξη θα είναι σημαντική και αυτό ακριβώς θέλω και εγώ να προσφέρω. Και θα έχω πολλά να πω ε, για το πώς έχουμε πάει μέχρι τώρα και για το τι θα κάνουμε στο μέλλον και εγώ και η, ε, μετά από μένα στο ίδιο αξίωμα. Αναφερθήκατε στο τι συνέβη ε, στη Βεγγάζη, κυρία Γκόμες, με τον Αμερικανό πρέσβη. Δεν θα σας εκπλήσει το να σα πω ότι στη συνάντησή μας και στο ταξίδι μας με την κυρία Κλίντον την περασμένη εβδομάδα ασχοληθήκαμε με το θέμα της Λιβύη και το τι μπορούμε να κάνουμε. Κάτι ε, το οποίο ο, Άμ μόλις ε, εκλεγής πρόεδρος των ΗΠΑ σίγουρα θα ε, είναι κάτι το οποίο θα απασχολήσει τον μόλις εκλεγέντα πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Και σίγουρα έχετε δίκιο ότι ε, το Μάλι έχει σχέση με, τις, ε, με την κατάσταση στη Λιβύα. Υπάρχει κάποια διακίνηση όπλων στο βορρά του Μαλί και αυτό από μόνο του έχει δημιουργήσει μια δυναμική που έχει κινητοποιήσει διάφορες ομάδες για πολλούς λόγους. Υπάρχουν πολλοί που είναι φονταμενταλιστές, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι είναι εγκληματίε, εμποροί ναρκωτικών. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι θέλουν ε, ένα διαφορετικό μέλλον. Υπάρχουν ε, πολλά και διαφορετικά κίνητρα για τις διάφορε ομάδες που δρούν εκεί. Και τα κράτη-μέλη κατανοούν ότι πρέπει από κοινού να δράσουν, πρέπει να συνεργαστούμε για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Ε, ιδιαίτερα στη Λιβύη που η αναμονή μιας κυβέρνησης για όλους μας ήταν μια δύσκολη κατάσταση και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε συνομιλητές επιτόπου. Ελπίζω ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε τα προγράμματα που προετοιμάζουμε. Ολοκληρωμένη δράση, συνεργασία με τους εταίρους μας ε, και άμεση δράση ε, και στη Λιβύη και στο Μαλή και μέτρα για την διασφάλιση των συνόρων. Νομίζω ότι αυτά είναι όλα τα στοιχεία που θα οδηγήσουν σε ένα ασφαλέστερο περιβάλλον. Κυρία Νέιτς, ρωτήσατε για τη Ρωσία. Συνεργαζόμαστε, συνεργαστήκαμε με τη Ρωσία στο Τσάντ, παραδείγματο χάρη, και με τον Σεγγέη Λαυρόφ. Ε, ένα από τα θέματα που συζητάμε ε, είναι η συνεργασία της Ρωσίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε κάποια από τα θέματα που αποτελούν κοινό μας μέλημα και πιστεύω ότι πρέπει να καταβάλουμε μεγαλύτερη προσπάθεια για να μπορέσουμε να επιλύσουμε κάποια από αυτά τα ζητήματα όπου δεν είναι πολύ διαφορετικές, τουλάχιστον θεωρητικά, οι θέσεις της Ρωσίας από τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως την υπερνηστερία και το τι θα κάνουμε στη, ε, στην περιοχή, με τους λαούς της περιοχής. Για την υπόθεση Μαγνίτσκι ε, και τι θα κάνουμε σε σχέση ε, με τις βίζες, υπάρχουν διάφορα θέματα στα οποία δεν συμφωνούν όλα τα κράτη-μέλη. Έχουμε θέσει αυτό το θέμα. Έχουμε στείλει μια επιστολή ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον πρόεδρο Πούτιν και θα συνεχίσουμε να ασχολούμεθα με το θέμα γιατί όπως είπατε είναι σημαντικό και υπάρχουν πολλά τα οποία πρέπει να κάνουν τα κράτη-μέλη. Οι συζητήσει ε, και η σχέση μας με τη Ρωσία θα είναι ένα ε, θέμα που θα έχει προτεραιότητα στην ημερήσια διάταξη, γιατί υπάρχει και η διάσκεψη κορυφής με την ε, Ρωσία, όπως γνωρίζετε. Κύριε Μπράντον, στο Μαλί, όπως είπατε και όπως γνωρίζουμε, υπάρχουν πολλέ ομάδε. Εγώ είχα πάει και στην Αλγερία και στο Μαρόκο και συζήτησα με του ανθρώπου επιτόπου για την περιφέρεια γενικότερα και για το τι μπορούμε να κάνουμε και τι άποψη έχουν οι ίδιοι. Είναι πολύ ενδιαφέρον ε, ε, ότι όσο ήμουν εκεί εξελισσόταν η κατάσταση. Τα μηνύματα τα οποία λαμβάναμε ήταν συνεχώς ε, καινούρια. Πρέπει να προσπαθήσουμε να ασχοληθούμε με τον πολιτικό διάλογο για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τις θέσεις μας. Συνεργαζόμαστε με το ελεκτικό συνέδριο ε, σχετικά με την ULEX. Θεώρησε ότι υπάρχει ένα σημείο στο οποίο δεν υπήρχε απόλυτη ισορροπία και πρέπει να δούμε τι δυνατότητα θα υπήρχε για να ε, βοηθήσουμε την κυβέρνηση στο Κωσυφοπαίδιο αντί ε, να προσπαθούμε εμείς να είμαστε πάντοτε παρόντες επιτόπου στο Νότο. Θέλουμε να υπάρχουν οι σωστοί άνθρωποι ε, τα κατάλληλα σημεία για να μπορούν να θέτουν αυτά τα θέματα. Οι διάφορε εκθέσει είναι ευπρόσδεκτε. Μερικέ φορέ δεν είναι τόσο ευανάγνωστε, αλλά είναι ευπρόσδεκτε διότι μα δίνουν μια εικόνα του τι φαίνεται ότι πρέπει να γίνει ε, από μια εξωτερική ματιά. Δεν συμφωνώ πάντοτε με όλα όσα περιλαμβάνονται στι εκθέσει, αλλά είναι χρήσιμο. Και ευχαριστώ πολύ για αυτό το οποίο είπατε για τον προπολογισμό. Θέλουμε να έχουμε μια ασφαλή γειτονία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουμε να εγγυηθούμε ισχυρή, ε, ειρηνική και οικονομικά ισχυρή ζωή για τους ανθρώπους επιτόπου. Κυρία Λόζινγκ, Ρωτήσατε για το Βόρειο Μαλί και αν συμφωνώ με αυτό το οποίο είπε ο ε, Γερμανός ε, αρχηγός του επιτελείου. Δεν ε, γνωρίζω επαρκώς τις λεπτομέρειες αυτών που είπε στα σχόλιά του. Αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι στο Μαλί έχουμε ακόμη πολλά να κάνουμε για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε περαιτέρω το έργο μας. Καταρχήν πρέπει να δούμε πώς θα υποστηρίξουμε την ΕΚΟΒΑΣ και αυτά που προσπαθεί να κάνει στο Μαλί, να τους βοηθήσουμε στην εκπαίδευση, στην υποστήριξη, να τους βοηθήσουμε ε, να βοηθήσουν εκείνους που προσπαθούν να μπουν στον πολιτικό διάλογο, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο ούτως ή άλλως, και όπως έχουμε κάνει, ε, όπως έχουμε κάνει και για την ε, πολιτική υγεία, θέλουμε να, να αντιμετωπίσουμε ε, τα θέματα ε, ε, των ανθρώπων επιτόπου, όπως κάναμε στο Σαχέλ, μέσω της ασφάλειας και της σταθερότητας να φροντίσουμε και τα θέματα της επιστηστικής βοήθειας. Και ούτως ή άλλως χρειάζεται μεγαλύτερη συμμετοχή μας και πρέπει να το κάνουμε με τον δέοντα τρόπο. Και γι' αυτό θα συνεχίσουμε να έχουμε διαβουλεύσεις με τους εμπλεκομένους όσο το δυνατόν περισσότερο. Ε, κύριε Γιάννης, με ρωτήσατε αν θα ανέφερα κάτι για μία συγχώνευση που δεν έγινε. Η απάντησή μου είναι όχι. Κύριε Κοπά, ρωτήσατε σε σχέση με την εμπειρία της επίσκεψης στο Βόρειο Κόσοβο και αν θα πρέπει ε, ε, η αποστολή της ΚΠΑ να υποκραστήσει την K4. Νομίζω ότι είναι θετική η σχέση μεταξύ της K4 και της EULEX αυτό το οποίο δεν λένε είναι ότι ανησυχούν για τη δυνατότητά μας να παρέχουμε αστυνομική υποστήριξη στο Βόρειο Κόσοβο. Και αυτό είναι μια ανησυχία γιατί δεν έχουμε επαρκή δυνατότητες και προσπαθούμε να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να δώσουν πρόσθετους πόρους. Αυτό που ανησυχεί την K4 είναι ότι θα χρειαστεί να πάρουν τη θέση ε, αυτού που θεωρούν ότι είναι ε, αστυνομική αντίδραση και όχι στρατιωτική αντίδραση. Τούτου λεχθέντο θα κάνουμε ό,τι μπορούμε με τους πόρους που έχουμε διαθέσιμου. και οι σχέσεις που έχουμε επιτόπου είναι ισχυρές. Οι σχέσεις μεταξύ της ε, K4 και της EULEX είναι πολύ καλές τώρα διορίζεται νέος επικεφαλής της EULEX, μόλις ολοκληρώθηκαν οι συνεντεύξεις ε, και μία από τις ερωτήσεις που έθετε στις συνεντεύξεις είναι πώς θα συνεργαστούν στενά με την K4. Είναι πολύ σημαντική η σχέση και σίγουρα είναι ένα θέμα πόρων, όπως πολύ σωστά επισημαίνεται. Κύριε Κάστιν, εσείς ε, συνεχίσατε σε σχέση με το Κόσοβο και είπατε ότι χρειάζονται περισσότερες συναντήσεις. Εγώ συναντήθηκα με τον Αντιπρόεδρο όταν ήμουν στο Κόσοβο με την ε, ε, Υπουργό Εξωτερικών, τον είπα την κυρία Κλίντον, συναντηθήκαμε με μέλη των διαφόρων κομμάτων και αν η σημερινή συνάντηση μας οδηγήσει και κάπου παραπέρα, είναι πολλά αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν. Και αυτή τη συνάντηση των Πρωθυπουργών τη θεωρώ ένα από τα βήματα, ένα από τα πολλά βήματα που θα πρέπει να κάνουμε όλοι θα πρέπει να ε, αισθάνονται ότι έχουν την υποστήριξη και την αναγνώριση που χρειάζονται ως άτομα και ως ε, ε, ιστορία. Κύριε Τάνακ, δεν ξέρω ποιος θα είναι ο επόμενος Υπουργός Εξωτερικών, τον είπα. Υπάρχουν βέβαια κάποια ονόματα τα οποία συζητούνται. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι όλα τα ονόματα που συζητούνται είναι πρόσωπα τους οποίους ε, έχω την τιμή να γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Επομένως, όποιος και να είναι ο επόμενος ε, ε, επιλεγής από τον πρόεδρο Ομπάμα θα είναι θετικό. Πάντως η συνεργασία μου με τη Χίλαρη Κλίντον ήταν πάρα πολύ ευχάριστη. Είμαστε πολύ καλοί συνάδελφοι και όταν πρότεινα να κάνουμε αυτή την κοινή επίσκεψη την περασμένη εβδομάδα πραγματικά με χαροποίησε πάρα πολύ γιατί είναι κάτι το οποίο είναι πολύ θετικό όταν να μπορούμε ε, να εκφράζουμε ένα κοινό μήνυμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάντως θα μου λείψει η κυρία Κλίντον, αυτό έχω να πω. Κυρία Κλινιτσέκ, για το ελεγκτικό συνέδριο και πάλι. Νομίζω ότι εν μέρει απήντησε σε προηγούμενη ε, απάντηση. Είναι μια σημαντική έκθεση και πρέπει να εξετάσουμε κάποια από τα θέματα τα οποία θίγονται. Αρκετά από τα θέματα ήδη έχουν συζητηθεί γιατί η έκθεση συντάχθηκε πριν από την ανθεώρηση και οι αλλαγές που έγιναν έχουν ε, ε, αντιμετωπίσει ορισμένα από τα θέματα που αναφέρονται στην έκθεση. Αναφέρονται κάποια θέματα τα οποία δεν μπορώ να ε, έχω εγώ υπό τον ελεγχό μου. Εγώ προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ με τις δυνατότητες που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με το διάλογό μας προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα και να διευκολύνουμε την κατάσταση επιτόπου. Όσον αφορά τη συμμετοχή των γυναικών, βεβαίως, το έχω πει πολλές φορές, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σε όλα τα θέματα που μας απασχολούν και ιδιαίτερα στην κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας να συμμετέχουν και γυναίκες. Θέλουμε να υπάρχει ισορροπημένη συμμετοχή των δύο φίλων στις αποστολές. Δεν είναι πάντοτε εύκολο να το διασφαλίσουμε αυτό, αλλά είναι και αυτό το τμήμα του επιχειρησιακού μας σχεδιασμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ήσασταν ε, πολύ πιο πειθαρχημένοι από τη, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με την τήρηση του χρόνου. Σας ευχαριστώ για όσα μας είπατε. Ο κύριος Μπρόκ ε, τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Νταζόν που προεδρεύσατε σε αυτή την συνάντηση. Θα ευχαριστήσω όλους όσους ήρθαν από το Βερολίνο, ειδικά για τη συνάντηση σήμερα. Ευχαριστώ τον κύριο Νταζόν για την έκθεσή του που είναι ένα σημαντικό έγγραφο για την περαιτέρω συνεργασία μαζί σας, κυρία Άστον, και με το Συμβούλιο. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε την πολιτική άμυνας που θα πρέπει να μπει στην ημερήσια διάταξη σε υψηλή προτεραιότητα. Υπάρχουν, υπάρχουν πολλές συνέργειες, ακόμη και αν το δούμε από πλευρά εξοικονόμησης χρημάτων. Νομίζω και αυτό μπορούμε να το λάβουμε υπόψη μας και είναι κάτι που μπορούμε να συζητήσουμε και με τα Εθνικά Κοινοβούλια και με τις ε, προτάσεις ε, που κάνει ο κ. Ντανζόν νομίζω ότι θα προχωρήσουμε σε αυτό το διάλογο. Σας ευχαριστώ πολύ που αφιερώσατε σήμερα το χρόνο για να έρθετε εδώ για να κάνουμε αυτή τη ε, συζήτηση. Σας συναντάμε πολλές φορές στην Ολομέλη, αλλά μερικές φορές είναι χρήσιμο να έχουμε και σε τέτοια ομίγυρη χρήσιμες συναντήσεις. πολλές φορές σημαντικές συζητήσεις γίνονται σε μικρότερες ε, σε μικρότερους χώρους συναντήσεων του Κοινοβουλίου. Μπορούμε να συζητήσουμε πιο αποτελεσματικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εύχομαι καλή συνέχεια.